στα πρακτικά θα έχουν εγκριθεί μέχρι το τέλος συνεδρίασης. Έχει έρθει η ώρα για τις επερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 130β. Το θέμα είναι η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ναυπηγικής Βιομηχανίας. Ο συνάδελφος Γιάκοφτσιτς έχει το λόγο για 5 λεπτά. Ο ναυτιλιακός εξοπλισμός και η ναυπηγική βιομηχανία υπήρξαν για δεκαετίε από του σημαντικότερου και στρατηγική συμμαχία βιομηχανικού κλάδου, απασχολώντας περίπου 450.000 άτομα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντική αυτή η κλάδη τόσο από οικονομική όσο και από κοινωνική άποψη, γιατί παρέχουν ποιοτική απασχόληση σε μεγάλες επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συμβάλλουν στην περιφερειακή βιομηχανική υποδομή. Στην Ευρώπη υπάρχουν περίπου 150 μεγάλα ναυπηγεία, πολλά από τα οποία αναπτύσσουν ενεργό δραστηριότητα στην παγκόσμια αγορά, με μερίδιο αγοράς περίπου 6% όσον αφορά τη χωρητικότητα. Παρ' όλα αυτά, κύριε Επίτροπε, τα κράτη με ναυπηγική βιομηχανία στην Ευρώπη είναι πολύ αδύναμα για να αντιμετωπίσουν τις ανταγωνιστικές πιέσεις από την Ασία, ιδίως από την Κίνα και την Νότια Κορέα, που εφαρμόζουν στοχευμένες ε, εθνικές στρατηγικές για την αυπηγική τους ε, βιομηχανία. Με πολύ σημαντική υποστήριξη. Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας Leadership 2020, Ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για τη δημιουργία μια ολιστική σφαιρική στρατηγική για την ευρωπαϊκή ναυτιλιακή και ναυπηγική βιομηχανία, προκειμένου να υποστηριχθεί η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα, η οικονομική βιωσιμότητα και η ανάπτυξη αυτού του σημαντικού τομέα λαμβάνει η Επιτροπή συγκεκριμένα μέτρα για τη διατήρηση και την ενίσχυση των υψηλή τεχνολογία και υψηλή αξία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τη Ευρωπαϊκή Ναυπηγική Βιομηχανία. Διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαφή πολιτική και μέτρα με στόχο την αντιμετώπιση του διεθνού αθέμητου ανταγωνισμού και τη έλλειψη κανόνων στο παγκόσμιο εμπόριο. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου, κύριε Επίτροπε. Πρώτα απ' όλα βέβαια θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ότι δεχτήκατε την πρωτοβουλία μου για, για τη διεξαγωγή συζήτηση για το θέμα αυτό και λυπάμαι που δεν ε, υπάρχουν άλλοι συμπατριώτες μου στην αίθουσα γιατί για την Κροατία η ναυπηγική βιομηχανία και η ναυτιλία είναι πολύ σημαντική κλάδη. Είναι γνωστό πόσο σημαντικό είναι να διαφυλάξουμε την επιβίωση της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας στην Κροατία κρατώντας και τις θέσεις απασχόλησης αλλά και την τεχνογνωσία και την εμπειρογνωμοσύνη γιατί το ναυπηγείο Ουλιάνικ στην Πούλα, στην Ίστρια, που γνωρίζω και καλύτερα, είναι πραγματικά φυτόριο ε, γνώσης, τεχνογνωσίες ε, και καινοτομία. Και θέλουμε μακροπρόθεσμη στρατηγική. Μαζί με το ναυπηγείο Ουλιάνικ και το ναυπηγείο της 3ης Μαΐου και το ναυπηγείο του Σπλίτ είναι σημαντικά ναυπηγεία που γνωρίζουν την ε, αγορά, αλλά χρειάζονται την ευρωπαϊκή και την εθνική υποστήριξη. Το μείζον πρόβλημα είναι κυρίως οικονομικό για τα ναυπηγεία. Η χρηματοδότηση της ναυπήγησης του πλοίου και η χρηματοδότηση του αγοραστή, του πλειοκτήτη. Γιατί αυτό κάνουν άλλε χώρε και αυτό είναι σημαντικό για να εξασφαλίσουμε την επιβίωση τη ναυπηγική βιομηχανία και όχι μόνο στην Κροατία. Θα ήθελα λοιπόν να παροτρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει συγκεκριμένου μηχανισμού και μέσα, ώστε με συγκεκριμένο και ανταγωνιστικό τρόπο να χρηματοδοτήσουμε την ναυπηγική βιομηχανία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πολύ, πολύ συχνά μιλούμε για την ανάγκη επαναβιομηχανοποίησης της Ευρώπης. Οπότε θα πρέπει να σώσουμε με αποτελεσματικά μέτρα ε, κάποιες βιομηχανίες που έχουν και οικονομική σημασία και τεχνικές γνώσεις για να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα στο μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας. Δεν θα πρέπει να διευκολύνεται η καθάριση των αυπηγείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να αποφύγουμε όμω κάτι τέτοιο, θα πρέπει να προσδιορίσουμε νέα μέτρα και κριτήρια, κάτι που μπορούν να κάνουν από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τι αρμόδιε αρχέ των ενδιαφερομένων χωρών μελών. Δεν μπορούμε με σταυρωμένα τα χέρια ε, να γινόμαστε μάρτυρε τη εξαφάνιση τόσο σημαντική οικονομική δραστηριότητα, ενώ οι εταίροι μα από άλλε περιοχέ του κόσμου ε, ασκούν τη δική του πολιτική και με επιχορηγήσει στηρίζουν τη δική του ναυπηγική βιομηχανία. Φυσικά θέλουμε ανοιχτή προσέγγιση ε, με γνώμονα την αγορά, γιατί και εγώ φιλελεύθερος είμαι, αλλά αν δεν είναι ελεύθερος ο ανταγωνισμός και είναι αθέμητος, πρέπει και εμείς να σώσουμε τη δική μας βιομηχανία, όπως κάνουν άλλες χώρες για τη δική τους. Και θα πρέπει να αυξήσουμε και το μερίδιο ε, της συναυπηγικής βιομηχανίας ε, στο παγκόσμιο εμπόριο. Γιατί τα ευρωπαϊκά πλοία, η ευρωπαϊκή ναυπηγική παραγωγή είναι σημαντική. Γιατί πολλές φορές ε, ναυπηγείται το πλοίο σε μία χώρα, αλλά από ανταλλακτικά και συστατικά μέρη που προέρχονται από διάφορα μέρη της Ευρώπης. Γι' αυτό ένας λόγος παραπάνω να διαφυλάξουμε το μέλλον της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Η Επίτροπο Μπιενκόφσκα έχει το λόγο εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσετε να συζητήσω ε, το θέμα αυτού του πολύ σημαντικού κλάδου της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Είναι πολύ σημαντικός κλάδος για τα περισσότερα κράτη-μέλη. Ε, θα αρχίσω ε, από το γενικότερο πλαίσιο Καθώς θυμάστε, τον περασμένο Σεπτέμβριο ο πρόεδρος Γιούνκερ έστειλε ένα πολύ έντονο πολιτικό μήνυμα για την ανάγκη ενίσχυσης τη βιομηχανία μα, έτσι ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική. Λίγες εβδομάδες μετά από αυτό παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την βιομηχανική πολιτική, η οποία εγκρίθηκε και περιείχε νέες ε, στρατηγικές, νέα σχέδια δράσης που θα καλύψουν τα κενά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έχουν ακόμα χρόνο για να ε, προχωρήσουν το θέμα, ακόμα και αν ε, δεν έχουμε πολύ από αυτό το χρόνο. Η βιομηχανική στρατηγική μας είναι οριζόντια, καλύπτει όλους τους τομείς, στόχο έχει την καινοτομία και την προσαρμογή, αλλά εντός του υφιστάμενου πλαισίου ο τομέας της ε, ναυπηγικής βιομηχανία είναι ένας μόνο από τους ε, τομείς τους οποίους εστιάζουμε. Βέβαια έχει πολλές ε, συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες. Επίσης λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα για στήριξη της, των αλλαγών και αυτό είναι ένα παράδειγμα του τι ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε. Ο ναυτιλιακός εξοπλισμός και η ναυπηγική πηγική βιομηχανία είναι πάρα πολύ σημαντικά οικονομικά. Έχετε πολύ δίκιο αγαπητέ συνάδελφε, διότι παρέχουν ε, θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη ε, των ε, χωρών και των εταιριών σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια της στρατηγικής leadership 2020 η πρωτοβουλία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική διότι δίνει έμφαση στην καινοτομία, στις δεξιότητες, στην χρηματοδότηση και στην στήριξη των ε, ναυπηγείων και της βιομηχανίας ναυτιλιακού εξοπλισμού. Όλες αυτές είναι προτεραιότητες ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά την πρώτη ερώτηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί προσπαθεί να στηρίξει την βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Η στρατηγική για το 2020 περιέχει ένα σχέδιο δράση. Οι περισσότερε επιμέρους δράσεις θα αναλυφθούν και θα εγκριθούν από τους ίδιου τους ενδιαφερόμενους φορείς. Βέβαια δεν επαναπαυόμαστε σε αυτό, αλλά κάνουμε και εμείς ε, από τη μεριά μας αυτά που μπορούμε. Τώρα η τρίτη φορής είναι ευπρόσδεκτη για να έλθουν σε εμά έτσι ώστε να συνεχίσουμε τα μέτρα. Προσπαθούμε να στηρίξουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ε, ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ευρώπη. Στα πλαίσια της άσκησης ε, Leadership 2020 ήταν να διερευνηθούν νέες ευκαιρίες ε, όσον αφορά το πρασίνισμα, τη διαφοροποίηση, το άνοιγμα σε νέες αγορές και την καινοτομία. Να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει μια πρόσφατη ιστορική απόφαση από την ναυπηγική βιομηχανία να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Είναι πρώτη φορά και είναι μια μεγάλη ευκαιρία για όλους. Στα πλαίσια της ε, στρατηγικής δίνεται έμφαση στην καινοτομία και ε, στις πράσινες τεχνολογίες. Και επίσης στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής θα έχουμε τη δυνατότητα να εξερευνήσουμε νέες δυνατότητες ε, της αγοράς, νέες ευκαιρίες και οχήματα και σκάφη που θα είναι ενεργειακά αποδοτικά. Ο ναυπηγικός τομείας δεν μπορεί φυσικά να επιβιώσει εάν δεν στηρίξουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο, την τεχνογνωσία και τις ε, σχετικές δεξιότητες. Έτσι λοιπόν το 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση της ε, ναυτιλιακής βιομηχανίας να δημιουργηθεί και να συσταθεί μάλλον ένα συμβούλιο για την ναυτιλία, στόχος του οποίου είναι να ε, δώσει έμφαση στην τεχνολογία και να διερευνήσει τις δυνατότητες ε, επέκτασης αυτής και καινοτομίες. Η τεχνολογία στον τομέα της ναυτιλίας έχει γίνει πάρα πολύ σημαντική, καθώς και η συνεργασία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων. Έχουμε επιλέξει λοιπόν κάποιους τομείς, 7-8 περίπου, μεταξύ των οποίων και ε, η ναυτιλία, που, θα, που συμπεριλήφθηκαν στην Ατζέντα 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στηρίζουμε διάφορα έργα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη ναυτιλιακής τεχνολογίας και με τη μορφή χρηματοδότησης. Μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, δηλαδή το 2018, ξεκίνησε η εφαρμογή της στρατηγικής αυτής. Σαφώς χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα και μία ξεκάθαρη στρατηγική. Όμως επιτρέψτε μου να ε, πω ότι πολύ σωστά μεν ε, αναφέρεται ότι η ναυτιλία και οι ναυπηγικοί στην Ευρώπη είναι, υστερούν σε σχέση με τον ανταγωνισμό από την Κίνα, όμως αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει στα πλαίσια της ομάδας εργασίας του ΟΣΑ για την ναυπηγική να ε, αναπτύσσει τον διάλογο με την Κίνα. Ε, ο στόχος ήταν να αναπτυχθούν σε ευκαιρίες για την Ευρώπη, να περιοριστεί η επιρροή και η επέκταση της Κίνας ε, στον τομέα αυτό στην Ευρώπη. Φυσικά αυτές οι, σχέ, αυτές οι προσπάθειες δεν έχουν άμεσα αποτελέσματα, είναι όμως ο μόνος τρόπος για να δείξουμε όχι μόνο στην Κίνα αλλά και σε όλους τα αμοιβαία ωφέλη της ε, σωστής συνεργασίας. Μετά, άμεσες επενδύσεις. Ε, σίγουρα η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ανοιχτή στις άμεσες ξένες επενδύσεις. Ας μην είμαστε όμως αφελείς. Αυτές οι άμεσες ξένες επενδύσεις δεν πρέπει να προσελκύουν επενδυτές οι οποίοι έχουν συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα προσπαθήσουν να εφαρμόσουν. Και φυσικά πρέπει ύψιστη προτεραιότητα να είναι η δημόσια τάξη και ασφάλεια και το Συμβούλιο και εμείς και ελπίζω και εσείς που θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό μέσω του ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων που ενέχουν κινδύνους των παράνομων εισαγωγών. Και τα ναυπηγεία συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο δράσης. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται μέσω διαφόρων μέτρων όχι μόνο να εντοπίσει τις προκλήσεις που έχουμε, αλλά να διατυπώσει συγκεκριμένες συστάσεις και να ανοίξει διάλογο με τους ε, ενδιαφερόμενους φορείς της βιομηχανίας έτσι ώστε να, αποτελέσει, να, κομμάτι, ε, να αποτελέσουν εκείνα να στο κομμάτι της ε, συνέχειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μπενκόφσκα, ο κύριος Κέλλη έχει το λόγο για τρία λεπτά. Πρόεδρε, επίτροπε και οι 5-6 συνάδελφοι που είστε εδώ. Είναι μεγάλη μου χαρά που εκπροσωπώ εδώ το ΕΛΚΑ σήμερα το απόγευμα. βεβαίω το ΕΛΚ είναι προσιλωμένο στη βιομηχανοποίηση τη Ευρώπη και στη διατήρηση τη ανταγωνιστικότητά μα. Θέλω να συγχαρώ και να επαναλάβω το ερώτημα της ομάδας ALDE για το θέμα τη ε, ναυπηγική βιομηχανία, το οποίο τόσο ωραία εξέθεσε ο συνάδελφο Γιάνκοβιτ. Το μέλλον του ευρωπαϊκού τομέα των ναυπηγείων ε, ε, κινδυνεύει και μόνο μια σαφής πολιτική που προσφέρει ενωμένη ε, και συντονισμένη προσέγγιση θα επιτρέψει στα ευρωπαϊκά ναυπηγεία να αντιμετωπίσουν τα, τις βιομηχανικές αλλά και κοινωνικές προκλήσεις. Θα πρέπει να μπορέσουμε να αντιπαρατεθούμε στους ε, ασιάτες ε, εταίρους μας. Η Ιρλανδία, η χώρα μου, είναι νησιωτική χώρα, γι' αυτό και έχει μια πολύ ζωντανή ναυπηγική βιομηχανία και θέλει να συμβάλλει στην ευρωπαϊκή προσπάθεια. Στις αρχές του, 20 και του, 1920 και του 1930 είχαμε το πιο σημαντικό ναυπηγεία στη χώρα, ε, το Harland and Wolff και εκεί απασχολούνταν 1.100 άνθρωποι. Πολλά μεγάλα σκάφη κατασκευάστηκαν ε, εκεί, όπως το Αλιάκνα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στον ναυτικό. Ε, δυστυχώς εκείνο το λιμάνι ε, έκλεισε το 1994 μετά από μεγάλες απώλειες και οδήγησε στην ε, συρρήκνωση. Το λιμάνι του Κόρκ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στον ε, χώρα που συμβάλλει ε, σημαντικά στις εξελίξεις. Μικρές τώρα ναυπηγικές μονάδες για την επισκευή πλοίων λειτουργούν ακόμα στο Κόρκ και σε ολόκληρη την Ιρλανδία. Το, επίσης το Λίμερικ στη δική μου περιφέρεια έχουμε, έχει ένα υπέροχο λιμάνι και τώρα ε, συνεργάζομαι με τον διευθυντή του, τον κύριο Κίτινγκ, είναι ένα από τα ε, φυσικά βαθιά λιμάνια της Ευρώπης και μάλιστα έγινε μια μεγάλη διάσκεψη στο Λίμερικ πρόσφατα ε, για τα λιμάνια και ευχαριστώ την Επιτροπή που συμμετείχε και επισκέφθηκε το λιμάνι. Έχουμε και πολλά μικρά αλευτικά λιμάνια στην περιφέρειά μου σε μέρη όπως το Κι και διάφορα άλλα μικρά λιμάνια. Είναι βασικά αλλιευτικά λιμάνια, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την οικονομία των ε, συγκεκριμένων ε, δήμων και κοινοτήτων. Έχουμε ακόμα το λιμάνι που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων. Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτό που είπε μια φορά ο Αντώνιο Ταγιάννη, να σταματήσουμε το βιομηχανικό σφαγιασμό της Ευρώπης και να βοηθήσουμε να αναζωογονηθεί η ναυπηγική μας βιομηχανία. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κέλλη. Ο κύριος Μάμικινς έχει το λόγο τώρα έχει μια ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να υποβάλω μια ερώτηση μέσω της γαλάζιας κάρτας. Η ναυπηγική βιομηχανία στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντική. Όμως ε, η Κίνα αποτελεί μεγάλο ανταγωνισμό στον τομέα αυτών. Θεωρείτε πως στο άμεσο μέλλον η Ευρώπη θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστική απέναντι στην Κίνα. Σας ευχαριστώ. Όχι μόνο θα είναι, αλλά οφείλει να είναι ανταγωνιστική. Και με εμψύχωσαν τα λόγια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα μέτρα που στοχοέχουν την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητάς μας και την υποστήριξη των λιμανιών μας. Θα πρέπει λοιπόν να, να να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας και έτσι πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ναυτική βιομηχανία να ανταγωνιστική την Κίνα και την ε, Νότια Κορέα και άλλες ε, χώρες. Γιατί, όπως είπα, ε, αυτό δήλωσε και ο Αντώνιο Ταγιάννη και πιστεύω ότι αν συνεργαστούμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τα κράτη-μέλη θα το καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κέλλη. Για πέντε λεπτά το λόγο έχει ο κύριος Μάμικινς. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι σημαντικός παράγων στην παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία, παρόλο που ε, μεγάλη ζήτηση αναμένεται στην παραγωγή την επόμενη δεκαετία, ε, που σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις ο κλάδος. Από ό,τι ε, βλέπω, ελάχιστοι έχουμε μείνει εδώ στη Ρολομέλη για τη συζήτηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το θέμα δεν είναι σημαντικό. Η Ευρώπη είναι μια ναυτιλιακή δύναμη και θα πρέπει να δούμε τι πλονεκτήματα και τι προοπτικές έχει ο κλάδος. Το ευρωπαϊκό μας σχέδιο είναι μοναδικό και αυτό θα πρέπει να ε, διαρωτηθούμε πώς θα εξασφαλίσουμε στα θέσεις κανονιστικό πλαίσιο. Ας μην ξεχνούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο κανόνες ε, και διατάξεις, είναι και γεωπολιτική στρατηγική. Και μάλιστα η ναυτιλία ε, είναι σημαντικό στοιχείο της πολιτικής της εξουσίας και για να είμαστε για πολιτική σημαντική παίκτη, θα πρέπει να προσέξουμε την αυτιλία μα. Η μελέτη που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Balance Technology Consulting δείχνει ότι η ευημερία του κλάδου τη ναυτιλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συμβάλλει όχι μόνο στην οικονομική και την πολιτική ασφάλεια, αλλά έχει και περιβαλλοντικέ επιπτώσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και σήμερα η Ευρώπη χρειάζεται μια ρεαλιστική και οραματική προσέγγιση στην αφηγική βιομηχανία. Και μάλιστα πρόσφατα έχουμε λάβει την απόφαση να συγκεντρώσουμε ε, την παραγωγή σε συγκεκριμένα ναυπηγεία υψηλής τεχνολογίας και η υψηλή τεχνολογία θα μας δώσει ανταγωνιστικό αποτέλεσμα ώστε να περάσουμε από το παρελθόν στο μέλλον. Ας μην ξεχνούμε όμως ότι και η Κίνα έχει τον πολιτικό στόχο της εισαγωγής στην ε, ναυπηγική υψηλής τεχνολογίας. Οπότε θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα για να διαφυλάξουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Από τη στιγμή που δεν έχουμε σαφείς εμπορικούς κανόνες παγκοσμίω, θέλουμε ε, ευρωπαϊκές διατάξεις για να προστατεύσουμε τους ναυπηγούς μας που αρχίζουν και δεινοπαθούν. Γιατί η, αγορά, παγκόσμια αγορά στηρίζεται στο δολάριο, οπότε θα πρέπει να προστατεύσουμε τη βιομηχανία από ε, χρηματοπιστωτικές ανισορροπίες και να έχουμε η συμμεταχείριση των παραγωγών. Επίσης, τα ναυπηγεία μας συμβάλλουν και στην ασφάλεια της ναυτιλιακής μας πολιτικής, στην πολιτική για την Αρκτική. Και σίγουρα τα κράτη-μέλη έχουν ισχυρά γεωστρατηγικά και ναυτιλιακά συμφέροντα. Και τα κράτη αυτά απρόθυμα θα εκχωρούσαν αρμοδιότητές του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν όμως πρέπει να ανταγωνιστούμε σημαντικές παγκόσμιες ναυτιλιακές δυνάμεις, θα πρέπει να συσπυρώσουμε και να συγκεντρώσουμε τους πόρους μας και να έχουμε κοινέ δράσεις. Έτσι θα ενισχύσουμε την ναυτιλιακή μας δύναμη και θα μας ε, επιτρέψει να δημιουργήσουμε μια κοινή ναυτιλιακή πολιτική. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια αποτελεσματική ε, ναυτιλιακή στρατηγική με περιβαλλοντικό προβληματισμό. Γιατί είμαστε η πιο προοδευτική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Και θα πρέπει τα κριτήρια αυτά να λαμβάνονται και στις ε, εμπορικές και ναυτιλιακές τις σχέσεις, ε, προκειμένου να προωθήσουμε τα υψηλά ε, περιβαλλοντικά μας πρότυπα. Επίσης και οι κλιματικές αλλαγές επηρεάζει τους κανόνες στην Αρκτική ειδικά και σε άλλες περιοχές και Ιδιαίτερα σήμερα που τα πλοία περνάνε περισσότερο από τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Ασία. Γιατί οι δρόμοι αυτοί θα είναι όλο και πιο επικίνδυνοι και θα μετα... Θα μετα... και γι' αυτό θα στραφεί ο ανταγωνισμό προ το βορρά, προ την αρκτική περιοχή. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε νέε τεχνολογίε με νέα πλοία που θα μπορούν ε, να πλέουν σε, κανό... σε συνθήκες ε, αντίξωε ε, ναυσιπλοείας. Στη Λετωνία η βασική πρόκληση της ναυπηγικής μας βιομηχανίας είναι να αναπτύξουμε νέες δεξιότητες και να προσαρμοστούμε στο σύστημα της αγοράς. Χάρη στους ιστορικούς κανόνες και τις παραδόσεις, η Λετωνία διατηρεί μια αξιοσέβαστη θέση στη, στη παγκόσμια ναυτιλιακή σκηνή. Και μάλιστα έχουμε νέες τεχνολογίες ε, Κατασκευή, νέο σχεδιασμό και πολλές καινοτομίε που δεν αρκούν όμως για να εξασφαλίσουν την οικονομική ευρωστία της λετωνικής ναυπηγική βιομηχανίας, δεδομένη τη μείωσης της ζήτησης στην Ευρώπη. Σίγουρα ε, ο κλάδος αυτός στηρίζεται σε μια τεχνολογία και η οικονομία της γνώσης και θέλουμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή προσέγγιση για να εξασφαλίσουμε την περαιτέρω ανάπτυξη της ναυπηγικής βιομηχανίας και την ευημερία των εργαζομένων σε αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ συναδελφέ κύριε Μάμικιν. Ακολουθεί η κυρία Κρούπα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, συμφωνώ απόλυτα με την προφορική ερώτηση του κυρίου Γιακόφτση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Κλάδο τη Ναυτιλία και τη Ναυπηγική Βιομηχανία. Ε, πολλό δε μάλλον που κάποιες προσωρινές δράσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είχαν κάποιες αρνητικές συνέπειες γιατί ξέρετε ότι η ε, γεννήθηκε στο Κντάνσκ τη δεκαετία του 70. Είχαμε χιλιάδες πλοία που ναυπηγήθηκαν εκεί. Δεν θα πρέπει λοιπόν ε, να κλείσουν αυτά τα ναυπηγεία. Θα θέλουμε συγκεκριμένες διατάξεις ώστε να μην χρειάζεται η υποστήριξη με δημόσια κονδύλια, με μια σωστή ιδιωτικοποίηση και να μην χαθούν ε, ε, εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. Χρειάζεται μια ε, διαδικασία αναδιάρθρωσης που δεν θα πρέπει όμως να οδηγήσει σε εξαγορά ή ε, εκποίηση μάλλον του ναυπηγείων του Γκτάνσκ. Μια ουκρανική ε, τελικά επιχείρηση αγόρασε τα ναυπηγεία του Γκτάνσκ και η συστηματική προσπάθεια εξουδετέρωσης των ναυπηγείων της ναυπηγικής βιομηχανίας τα τελευταία 30 χρόνια είναι απαράδεκτη. Δεν θα πρέπει να έχουμε τέτοια φαινόμενα στην Ευρώπη. Ε, έχουμε στο Στέτσιν, στο Κτάνς και στο Κδίνια σημαντική ναυπηγική βιομηχανία που μάλιστα έχει στρατηγική σημασία για την ασφάλεια της κάθε χώρας και την καταπολέμηση ε, των απειλών που δημιουργεί ο αθέμητος ανταγωνισμός από τρίτες χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκρούπα. Για τρία λεπτά η κυρία Άντερσον έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Η Ιρλανδία είναι ένα νησί και ω νησί εξαρτάται περισσότερο από την ναυτιλία από τα περισσότερα κράτη-μέλη. Η συνεχής όμως απερισκεψία τη βρετανική κυβέρνηση ως προς τον Brexit σημαίνει ότι είναι πολύ συνετό να αυξήσουμε την ναυτιλιακή μας ικανότητα προκειμένου να αποφύγουμε να τιμωρηθεί η Ιρλανδία από τι πιθανέ δυσκολίε που θα έχουν στη μετακόμιση των Ιρλανδικών εξαγωγών μέσω τη Βρετανία στα εμπορεύματα. Οπότε η ναυτιλία και η ναυπηγική βιομηχανία αποκτούν αυξανόμενη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την αντιμετώπιση τη οικονομική κρίση στο ναυπηγείο ε, ε, υποστηρίχθηκε από το ναυπηγείο Χάρλαντ και Βόλφ, που είναι το σημαντικότερο ναυπηγείο στην Ιρλανδία και βρίσκεται στο Μπέλφαστ. Έχουν κάνει ένα άνοιγμα προ την τεχνολογία και την καινοτομία. Είναι όλο και πιο ε, οικολογικά προσανατολισμένο αυτό το ναυπηγείο και διαφοροποιείται προ νέε αγορέ. Πολλά εξαρτώνται από το ναυπηγείο αυτό και ε, τα λιμάνια του, βορρά, του Βορρά, κυρίως το Belfast, το Warren Point, το Λάρν και ε, της μου του Foil Port που θέλουν σύνδεση με την ευρωπαϊκή αγορά και εξαρτώνται και τα ε, λιμάνια αυτά από την ευρωπαϊκή αλυσίδα προμηθειών. Ενώ το Brexit θα πλήξει ανεπανόρθωτα αυτό το σχέδιο και μπορεί να οδηγήσει σε, σε μεγάλο πλήγμα στον κλάδο. Μάλιστα, η Βρετανική κυβέρνηση φαίνεται ότι στηρίζεται περισσότερο και εξαρτάται από τα κανονιοφόρα από το να έχει ένα συγκεκριμένο όραμα για τον κλάδο. Επίση, φαίνεται να ξεχνά η Βρετανική κυβέρνηση τι συνέπειε που θα έχει το Brexit για τη Βόρεια Ιρλανδία. Όλα αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο σχεδιασμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το μέλλον. Υπάρχουν κάποιε ε, λύσει για τι απειλέ που δημιουργεί το Brexit για τον κάθε κλάδο, συμπεριλαμβανομένε και τη ναυπηγική βιομηχανία. Έχουμε παρουσία παρουσιάσει αυτές τις λύσεις ε, ε, μέσω της πρώτης που κάναμε για ειδικό καθεστώ για τη Βόρεια Ιρλανδία και την παραμονή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον Brexit. Επίσης, ε, προτείναμε το σύστημα των πράσινων και κόκκινων διάβλων που συμπληρώνουν την υπάρχουσα υποδομή των λιμένων και θα μπορούσαν να εξυπηρετούν την εισαγωγή και εξαγωγή από τη Βόρεια Ιρλανδία των εμπορευμάτων. Ε, επίσης, ε, αυτό το σύστημα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τα διαμετακομιζόμενα αγαθά από τη Βρετανία προς τη και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, προασπίζει την ακαιρεότητα της ενιαίας αγοράς ε, και επιτρέπει την καλύτερη συνέχιση του εμπορίου από την Ανατολή προς τη Δύση. Δεν θέλουμε να ενισχυθεί ένα, το σκληρό σύνορο και να ξαναχωρήσει την ε, Ιρλανδία. Ούτε θέλουμε ένα θαλάσσιο σύνορο μεταξύ Βρετανίας και Ιρλανδίας. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι το πλοίο Τιτανικός ε, κατασκευάστηκε στο ναυπηγείο Χάρλαντ και Γουόλφ στο Μπέλφαστ. Ε, το κέντρο της, του Μπέλφαστ και η συνοικία του Τιτανικού, χάρη στην ειρηνευτική διαδικασία, αναπλάστηκαν και και είδαν πολύ θετικέ εξέλιξει. Θα πρέπει να σε υπενθυμίσω όμω ότι ο Τιτανικό στο παρθενικό του ταξίδι χτύπησε σε παγόβουνο στο Βόρειο Ατλαντικό και βυθίστηκε. Α μην αφήσουμε την Ιρλανδία, τη Βόρεια και τη Νότια να συντριβούν στο παγόβουνο του Brexit. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Άντερσον. Για τρία μισή λεπτά η κυρία Έλισεν έχει το λόγο. Ο κύριο Έλισεν. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ακόμα περισσότερη νομοθεσία για τον ε, ναυπηγικό τομέα. Δεν συμφωνούμε με αυτά τα σχέδια, κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούμε πως ε, παρεμβαίνει. Παρεμβαίνει με τρόπο παράλογο ή υπάρχει υπερβολική νομοθεσία. Εμείς είμαστε υπέρ μιας ε, οικονομίας της ελεύθερης αγοράς, όπου οι επιχειρήσει είναι υπεύθυνε για την επιτυχία τους ή την αποτυχία τους. Ε, οι γραφειοκράτες δεν έχουν ε, εικόνα της κατάστασης, δεν ξέρουν τι σημαίνει υγιή ανταγωνισμός και ελεύθερη αγορά. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε κατά της μεταφοράς αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά της κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος και κατά της διάσωσης ναυπηγείων τα οποία οδεύουν προς την καταστροφή. Πιστεύουμε πως η χρεοκοπία απλά θα παραταθεί, δεν θα αποφευχθεί. Ας ε, δούμε το αν τομέα της αεροναυπηγικής για παράδειγμα ή άλλους τομείς. Ε, βλέπουμε πως έχουν κατασπαταληθεί κονδύλια. Τη δεκαετία του 80 η κυβέρνηση της χώρας μου έδωσε εκατομμύρια για να διασώσει τα ναυπηγεία και δεν τα κατάφερε. Τα μεγάλα ναυπηγεία έκλεισαν και χάθηκαν χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. Όλα αυτά λοιπόν ε, δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Τα χρήματα των φορολογούμενων εξαφανίστηκαν, εξατμίστηκαν. Η αναβίωση ορισμένων κλάδων δεν έχει γίνει λόγω της κρατικής στήριξης, αλλά λόγω της επιχειρηματικότητας και της εφευρετικότητας των ίδιων των επιχειρήσεων. Η ίδια η αγορά είναι αυτή που θα αποφασίσει πού, πότε και πώς ε, θα υπάρχει ε, παραγωγή αγαθών. Έχει να κάνει με τους νόμους της προσφοράς και της ζήτηση. Γι' αυτό πρέπει να σταματήσουμε να επιχορηγούμε ε, τα πάντα, να ελέγχουμε τα πάντα και, να αφήσουμε, και πρέπει να αφήσουμε τον τομέα της ε, ναυπηγικής ομηχανίας στην ησυχία του. Σας ευχαριστώ πολύ. Για 3,5 λεπτά ο κύριος Τζαμπάτσκι έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Γιάκοφσιτς που έθιξε αυτό το τόσο σημαντικό ε, θέμα. Πολλά κράτη-μέλη έχουν ε, ναυπηγική βιομηχανία η οποία απειλείται. Γίνεται πολλής λόγος για την ε, εκ νέου βιομηχανοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται όμως να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης, να διατηρηθούν αυτές οι παραδόσεις. Ναι, είναι, υπάρχει ανταγωνισμός από πλευρά τρίτων χωρών που δεν είναι πάντα θεμητός, αλλά αυτό είναι απόλυτο φυσιολογικό. Είναι χώρες που θέλουν και αυτές να μπουν σε αυτήν την αγορά. Από εμά εξαρτάται, από τα κράτη, ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, να δούμε πώς θα διατηρήσουμε αυτές τις θέσεις απασχόλησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τζαμπάτσκι. Ο κύριος Μάμικινς έχει μια ερώτηση για εσάς. Κύριε Μάμικινς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τζαμπάτσκι, Ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε την ερώτησή μου. Η Λετωνία, η χώρα μου, το 2004 έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Βουλγαρία αργότερα, το 2007, μαζί με τη Ρουμανία. η δική μας ναυπική βιομηχανία έχασε τελικά. Όμως είχαμε και αρκετά ωφέλη τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις. Πώς, έγινε, πώς ήταν τα πράγματα στη χώρα σας, χάσατε, κερδίσατε, τι ακριβώς. Колега, благодаря за въпроса, колега Мамикинс. Вие сте прав, влизането в Европейския съюз, както на Латвия, така и на България, въпрос... Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Είναι θέμα διαπραγμάτευση ε, για τη Λετωνία και την Βουλγαρία. Ναι, αρχικά χάσαμε πολλέ θέσει απασχόληση, αλλά στη συνέχεια αναπτύχθηκε αυτό ο τομέα. Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο δημόσια ναυπηγεία και πολλά ιδιωτικά. Οπότε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνεργαστούμε μεταξύ μας για να, ε, ε, και στον τομέα της ναυτιλίας για να μπορέσουμε να έχουμε πιο θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τζαμπάτσκι. Δεν υπάρχει κάποιο συνάδελφο που θέλει το λόγο στη διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑ. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσω το λόγο στην κυρία Πινκόσκα για να κλείσει την ε, συζήτηση. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ όλου εσά για τα σχόλιά σα. ήθελα να πω ότι η ναυτιλία και η ναυπηγική βιομηχανία είναι πάρα πολύ σημαντική σε βιομηχανίε και χρειάζονται ακόμα περισσότερε δράσει από αυτέ που γίνονται τώρα για του επόμενου 18 μήνε. Όπω ανέφερα ήδη, το πρόγραμμα Leadership 2020 αποτελεί ένα πλαίσιο που θα δώσει τον ε, κατάλληλο προσανατολισμό έτσι ώστε να ενστερνιστούν επιχειρήσει στις νέε ευκαιρίε και να ε, προχωρήσουν στην ψηφιοποίηση, στι νέε τεχνολογίε ε, κτλ. Είμαι σίγουρη πως ε, φυσικά θα υπάρχει κάποια καθυστέρηση, διότι αυτό συμβαίνει σε ένα διάλογο που συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Θεωρώ όμως ότι θα συνεχίσει αυτός ο διάλογος να δίνει τα κατάλληλα αποτελέσματα στο μέλλον. Φυσικά αρκετά κράτη-μέλη φροντίζουν έτσι ώστε η ναυτιλία και η ναυπηγική να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος και στις ευκαιρίες που προκύπτουν. Και φυσικά συνεχίζουμε τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη, με τους ενδιαφερόμενους φορείς, με εκπροσώπους της βιομηχανίας, όμως να είστε σίγουρος ότι θα συνεχίσω να δίνω μεγάλη προσοχή σε τομείς ε, όπου θεωρώ πως πρέπει να εντείνουμε τις ε, δραστηριότητές μας και σε τομείς όπου μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση, για παράδειγμα, πρόσβαση στην αγορά. Ε, λαμβάνονται πολλά μέτρα για τις δεξιότητες, για την πρόσβαση σε νέες αγορές, όμως θεωρώ πως θα έχουμε καλά ε, νέα και πως θα έχουμε θετικά αποτελέσματα όταν θα συζητήσουμε το θέμα του προπολογισμού. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα περιμένουμε να δούμε μέχρι τότε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Επίτροπε.